Okay, um, Προτείνω να συνεχίσουμε με τις εργασίες μας ε, στην ΙΜΚΟ και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης για το ε, σχέδιο για την ε, στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο. Είναι μια γνωμοδότηση της ΙΜΚΟ, ΙΝΤΑ και Νομικής Επιτροπής και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ντάλτον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την γνωμοδότηση της ΙΜΚΟ. Θα ήθελα να ασχοληθούμε με τον αντίκτυπο πάνω ε, στους ε, καταναλωτές ε, για να δούμε τις λήψεις και τις σχέσεις με το εμπόριο. Πρώτον, για το ηλεκτρονικό εμπόριο, νομίζω ότι αυτό με αυτό ασχολούνται ε, οι καταναλωτές, έχουμε την στρατηγική για μέσα στην ψηφιακή αγορά, έχουμε τον γεω αποκλεισμό, το χάρη αν επιληθεί το θέμα, ε, θα μπορέσει η στρατηγική αυτή να ανθίσει. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εμπόριο που ευημορεί μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η διευκόλυνσή της του δεν έχει βελτιωθεί. Και οι καταναλωτές πολύ συχνά έχουν όταν ε, προσπαθούν να αγοράσουν κάτι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν ιστότοπο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ συχνά ε, ε, κάποιο, κάποιος τους χτυπάει την πόρτα ή λαμβάνουν ένα γράμμα με πρόστιμα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, ιδαλλιώς δεν θα έχουμε την ηλεκτρονικό εμπόριο να ευημερεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, εγώ ε, ε, μιλάω για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτό ισχύει και για άλλα, άλλες χώρες. Αν αγοράσετε κάποιον, θα έχετε έναν δασμό αν 135 λιρών και επίσης ΦΠΑ εισαγωγικό 15 λίρες, 17 ή 18 ευρώ δηλαδή. Βεβαίως, ε, έχει ορισμένα δικαιώματα αγοράς ένας ε, ταξιδιώτης 390 ε, λιρών μπορεί να αγοράσει όταν εισάγεται στη χώρα και δεν έχει εισαγωγικούς δασμούς και δεν χρειάζεται να δηλώσει τίποτα κάτω από αυτό το επίπεδο. Υπάρχει εδώ μια διαφορά ανάμεσα στα δύο. Μια, αν θέλουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο να ευημερεί παγκοσμίω, θα πρέπει να ρυθμίσουμε αυτή τη διαφορά. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που προσπάθησα να αντιμετωπίσω στην γνωμοδότηση. Πρέπει επίσης να το βάλουμε αυτό στο θεματολόγιο ε, του ΠΟΕ. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει ε, στην ημερήσια διάταξη στα πλαίσια μιας ένας ευρύτερου θέματος σχετικά με την, το ψηφιακό εμπόριο και τους φραγμούς που υπάρχουν. Έχουμε επίση στη ΣΤΑΜ την προστασία των καταναλωτών που είναι κάτι το σημαντικό για το εμπόριο, τα πληρωμές, η διαφάνεια ε, και πέραμπτος χάρη ε, για τα μέσα τα διαδικτυακά και λοιπά για διάφορα προϊόντα να μην υπάρχουν μεταχειρήσεις ε, που επιφέρουν διακρίσεις. Επίσης η ελεύθερη ροή και κυκλοφορία δεδομένων που είναι ένα επίκαιρο θέμα, αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο όλων και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, ε, ότι χρειάζεται καμιά φορά η ψηφιοποίηση για λόγους ασφαλείας, αλλά οι περιορισμοί της ροής δεδομένων μπορεί να είναι ένας προστατευτισμός συγκαλυμμένος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη ροή και κυκλοφορία δεδομένων. Αυτό λέγεται ότι δεν πρέπει να γίνεται σε συμφωνίες εμπορικές, το αναγνωρίζω αυτό. Η καλύτερη προσέγγιση για να εγγυηθούμε την ελεύθερη ροή είναι να προστατεύσουμε ε, την ε, τα κανόνες ε, προστασίας δεδομένων και ιδιωτικής ζωής που έχουμε αυτές ε, ε, να έχουμε συμφωνίες με διάφορες χώρες του κόσμου καταλληλότητας όπως με την Ιαπωνία θα πρέπει η Κομισιόν να εξετάσει αυτές τις συμφωνίες που υπάρχουν με άλλες χώρες του κόσμου και την προστασία των δεδομένων και ως αλλάζουν στο μέλλον αυτή θα πρέπει να αλλάξουμε με τις εμπορικές συμφωνίες. Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Επίσης έχουμε διάφορους φραγμούς οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι και δυσκολίες. Υπάρχουν τα NTB. Γιατί υπάρχουν NTB για μια μικρή χώρα. Αυτό νομίζω είναι μια δημόσια πολιτική και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση, αλλά είναι η ε, περίπτωση σχετικά ε, με την ψηφιακή κατάσταση. Χρειαζόμαστε να γίνει περισσότερη εργασία στο επίπεδο του ΠΟΕ για να εξαλείψουμε φραγμούς και εμπόδια και θα πρέπει να προωθήσουμε ε, ένα εργαστήριο παγκόσμιο σχετικά με τα ψηφιακά θέματα, σχετικά με την στρατηγική πρόοδος έχει ε, γίνει ε, και νομίζω ότι έχουμε ένα πλαίσιο φιλικό προς τον καταναλωτή τον 21ο αιώνα. Θα ήθελα οι συνάδελφοι να πούνε ε, τις απόψεις τους, συνεργάζομαι με τους κοιόδης εισηγητές στενά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ σκιώδης, είναι ε, ο κύριος Πόσπης, δεν τον βλέπω όμω. δεν ξέρω ποιο άλλο είναι κανένα από το ΕΛΚ, όχι. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, η κυρία Γκέριγκερ Ντεόντεμπερ, απούσα επίση. και κανείς δεν την αντικαθιστά. Um, so, um, we go then... Και θα περάσουμε αμέσως στον κύριο Άλμπρεχτ, εξ ονόματο των Πρεσίνων. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να έχουμε ε, μαζί τους συναδέλφους ε, όταν θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης. Προσβλέπω στη συζήτηση αυτή, βεβαίω με ενδιαφέρει πάρα πολύ και όλα αυτά που είπε ο κύριος Ντάλτον με ενδιαφέρουν για την ε, διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και στις περιβαλλοντικές. Βεβαίως, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μην χάσουμε τη δυνατότητα πίεσης ε, στους ε, εμπορικούς μας εταίρους να αυξήσουν την προστασία προσωπικών δεδομένων στην τάξη τους. Και πιστεύω ακράδαντα ότι και αυτές οι αποφάσεις ε, στο νέο κανονισμό θα είναι καθοριστικές. Αυτός είναι ο βασικός μας σύμμαχος ή ε, δρόμος. Αλλά έχουμε και άλλες δυνατότητες. Αλλά δεν θα πρέπει να πλατιάζουμε πάρα πολύ και να διευρύνουμε την ανάγκη βεβαίως καταπολέμησης των επιθετικών εμπορικών πρακτικών. Δηλαδή, να μην έχουμε καταχρηστικά τέλη και εμπορικούς φραγμούς. και αθέμητες διατάξεις εντοπισμού των δεδομένων. Πολλές είναι και άδικες. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για την απρόσκοπτη ροή των δεδομένων. Δεν είναι μόνο τα προσωπικά δεδομένα, υπάρχουν και άλλες ε, καταστάσεις, όπως π.χ. κάποια ζητήματα πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων που μπορεί να ανακύπτουν. Άρα, δεν θα ήταν φρόνιμο να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτη ροή και τελείωσε και εμεί θα πρέπει να διαπραγματευτούμε κάποια πρότυπα και προδιαγραφές. Ελπίζω τελικά να είναι ισόρροπη η ε, γνωμοδότησή μας για τις διαπραγματεύσεις στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και να βρούμε ένα καλό τρόπο για να προστατεύσουμε και το δικό μας σύστημα ε, προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο συνάδελφο που να ζητά το λόγο για το θέμα αυτό, οπότε να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε την έκθεση και να επιβεβαιώσω ότι ήδη τα έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Και από τη δική μας πλευρά συμμεριζόμαστε τι τρεις αρχές από τον οποίων θα πρέπει να εδράζεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ανάγκη ε, εξυγχρονισμένων εμπορικών κανόνων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εμπορευμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ψηφιακή επανάσταση, τι εξελίξει στον χώρο τον ψηφιακό αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και ωφέλη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Από τη δική μας την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη απαντήσαμε στην ανάγκη αυτή με την κατάρτιση ενός κεφαλαίου για τα ψηφιακά θέματα στις διαπραγματεύσεις του χάρη με το Μεξικό με συγκεκριμένη ε, απαγόρευση για τελευνικούς δασμού στι ηλεκτρονικέ επικοινωνίες, για την ε, απαγόρευση και άλλων ε, πρακτικών Είμαστε πιο φιλόδοξοι από άλλου ε, διαπραγματευμένου. Επίση υπάρχουν ρήτρε για να συζητείτε η διαλογικότητα των προτύπων και άλλα ζητήματα που αναφέρονται και στην έκθεση. Επίση, εάν δούμε την πρόσφατη συμφωνία με την Ιαπωνία και τις αρχές που ακολουθήσαμε εκεί, νομίζω μπορούμε να το θεωρούμε ένα καλό ορόσημο στην όλη περιοχή, γιατί και εκεί υπήρξε ειδικό κεφάλαιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο ανταποκρίνεται στα βασικά αιτήματα, την πλειοψηφία των ε, ζητημάτων που αναφέρονται στο δικό σας κείμενο. Ένα θέμα που είναι σημαντικό και στο οποίο θέλω να σταθώ γιατί αναφέρθηκε και εδώ για τη ροή δεδομένων. Το θέμα είναι πραγματικά ε, ύψης της σημασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συζητήσεις εντός των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά για να πετύχουμε μια κατάλληλη ισορροπία από τη μια μεταξύ του να ε, προλάβουμε την αδικαιολόγητη ροή δεδομένων ενώ ταυτόχρονα να διατηρούμε και να διασφαλίζουμε τη δυνατότητα των ε, πολιτικών να ορίζουν την προστασία των δεδομένων. Θα πρέπει να μην <clears throat> πληγεί η ανεξαρτησία διπλωμάτευση ε, για εμπορικέ συμφωνίε, γι' αυτό συνεργαζόμαστε εδώ και με το Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά ένα παράδειγμα πάλι συμφωνία με την Ιαπωνία, πρόσφατο. Ε, υπάρχει η δυνατότητα λήψης αποφάσεων που μπορεί να έχουν πολύ θετικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε λοιπόν ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αναγνωριστεί στην έκθεση. Συνολικά, Στηρίζουμε λοιπόν την έκθεση, μπορούμε να συμφωνήσουμε δηλαδή, το φάσμα των θεμάτων που καλύπτονται, το γεγονό ότι στην ε, γνωμοδότηση περιλαμβάνονται συστάσει για τι διαπραγματεύσει των ΠΟΕ. Να θυμίσω ότι προσφάτω η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πρόταση για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που να διευκολύνονται οι επιγραμμικές συναλλαγές. Αυτό καλύπτει και συμπεριλαμβάνει κάποιες ε, ρήτρε και ιδιωτικέ διατάξεις όπως τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, την προστασία των καταναλωτών, το spam. Ε, όποτε συζητάμε τα θέματα αυτά, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε 164 μέλη και το επίπεδο των φιλοδοξιών ε, αυτομάτως ε, πέφτει. Πάντω, να μην ξεχνάμε ότι οι συζητήσει στον ΠΟΕ για το θέμα αυτό είναι δυσχερέστατε λόγω των αναπτυσσόμενων χωρών. Γι' αυτό χαιρόμαστε που βλέπουμε στην έκθεση την ειδική ε, μνήμα στι ιδιαίτερε αυτέ εξελίξει. Συνολικά, λοιπόν, συμφωνούμε με την κατεύθυνση τη δουλειά σα και ανυπομονούμε να συζητήσουμε περαιτέρω και να μελετήσουμε την έκθεση αυτή. Πολύ σα ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θέλει ο εισηγητή να προσθέσει κάτι. Ναι πολύ γρήγορα. Είναι πολύ εύκολο να διαπραγματεύεται κανεί όταν ε, υπάρχουν μόνο δύο ομάδε στην αίθουσα. Και νομίζω το θέμα δεν είναι πολύ αμφιλεγόμενο. Οι περισσότερε ομάδε μάλλον συμφωνούν. Στον κύριο Όλμπρεχτ να πω ότι τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά διαμακρών και δεν είναι πραγματικά αρμοδιότητα της ΣΥΜΚΟ. Και εδώ για την προστασία των καταναλωτών βεβαίω είναι αρμοδιότητα τη Επιτροπής μας. Και γι' αυτό τα συζητάμε εδώ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εντείνουμε κάπως τη δουλειά μας, αλλά δεν νομίζω ότι απέχουμε από το να βρούμε συμφωνία. μόνο και για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, και για τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Η προθεσμία για την υποπολίτη είναι στις 6 Σεπτεμβρίου. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή εξέταση των τροπολογιών στο σχέδιο γνωμοδότησης για την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τι διαδικασίε που υποστηρίζουν τι δημοπρατεύσει σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τη Ένωση στι αγορέ δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών. Πολύ μεγάλος ο τίτλος. Να δώσω το λόγο αμέσως στον εισηγητή για το θέμα αυτό, τον κύριο Στέφανετ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια πρώτη πρόταση για τον κανονισμό αυτό ήδη από το Μάρτιο του 2012 προκειμένου να καθορίσει το λεγόμενο εργαλείο ε, για της δημόσιας προμήθειας διεθνώς. Ο σκοπός είναι να ε, αυξηθεί η βαρύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, ώστε να υπάρχουν και περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης για τους Ευρωπαϊ... Ευρωπαίους ε, οικονομικούς σε αγορέ ε, δημόσιων προμηθειών τρίτων χωρών. Το Κοινοβούλιο είδε να έκτηνε τροπολογία στην πρόταση τον Ιανουάριο του 2014 και το θέμα αναπέμφθη στην Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό για να τα εξετάσει περαιτέρω. Ωστόσο το Συμβούλιο ήταν διχασμένο προς τη συγκεκριμένη πρόταση με ε, ίσο αριθμό κρατών μελών και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Δηλαδή κάποιοι επέκριναν και κάποιοι εξέφρασαν γενική υποστήριξη στην Ολυδέα. Το Συμβούλιο ε, ακόμη δεν έχει βρει λύση για το θέμα αυτό τώρα, οπότε το Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει ε, τριμερείς διαλόγους μαζί ε, Το σχέδιο αυτό γνωμοδοτησία συμπεριλαμβάνει τι τροπολογίε που είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή ΙΜΚΟ ήδη από, τον Οκτώβριο, ε, από τις 17 Οκτωβρίου 2013. Ε, στις διατάξεις που διατηρήξαμε ανέπαφε στην αναθεωρημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαμε κοινέ και αποκλειστικέ αρμοδιότητες τη ΙΜΚΟ και κάποια από τα σχόλια αυτά έχουν ε, χρησιμοποιηθεί και στι αναθεωρημένε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2016. Και χθε είχαμε μια συνάντηση σκιωδών ε, με του υπόλοιπου συναδέλφου και να ενημερώσω του ε, συναδέλφου εδώ ότι εγώ ζητώ να αποσυρθούν όλε οι τροπολογίε που άπτονται αρμοδιοτήτων τη ΙΜΚΟ. Θα καταλήξουμε σε συμβαστικέ τροπολογίε, ιδίω για τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, ούτω ή άλλως. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ και νομίζω ότι τόντι πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα και να περιοριστούμε στις δικές μας αρμοδιότητες. Θα συμφωνήσω. Ε, οπότε να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Γκραπίνη που είναι η σιώδη συζητήτρια για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Στέφανετς όπως είπε προτείναμε, είχαμε μάλλον συνάντηση σχεδόν χθε και νομίζω ότι καταλήξαμε σε μια συμβαστική λύση που είναι ικανοποιητική σε μεγάλο βαθμό. Οπότε, οι τροπολογίε που υποβάλαμε στις συνεδρίες των ε, σχεδόν θα πρέπει να είναι εντό του πεδίου των αρμοδιοτήτων μας. Γι' αυτό επιμείναμε σε τρεις τις διάβασα και τις ξαναδιάβασα. Είναι τροπολογίες των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Από τις 16 επιμένουμε σε 3 και μερικές από αυτές τις τροπολογίες άπονται των αρμοδιοτήτων μας. Ελπίζουμε λοιπόν να συμπεριληφθούν στις συμβαστικέ. Θέλω να τονίσω μετά από αυτήν την ε, εισήγηση του συναδέλφου ότι η έκθεση αυτή, η γνωμοδότηση αυτή ε, μας χρειάζεται. Γι' αυτό έθεσα σήμερα και τις σχετικές ερωτήσεις της Υπουργός, της, της Υπουργούς της Εστονίας. Το χρειαζόμαστε αυτό το νέο εργαλείο, γιατί θα δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πρόσβαση και να ανοίξει τις αγορές για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα των δημόσιων προμηθειών. Ε, και μάλιστα θα ασκήσει πίεση κατά του προστατευτισμού κάποιων χωρών. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή και σήμερα το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής εταιριών τρίτων χωρών με ένα τζίρο πολύ σημαντικό, 12 ευρώ. Υπάρχουν όμως τρίτα κράτη που από την πλευρά τους ε, έχουν τόσο αυστηρούς κανόνες που δεν επιτρέπουν σε χώρες ή σε εταιρείε δικές μας να συμμετάσχουν στις δημόσιες προμηθείες τους. Είναι λοιπόν σημαντικό το θέμα αυτό να ε, διευθετηθεί και θα πρέπει να υπάρξει και καλή επικοινωνία. Ε, δεν θέλουμε προστατευτισμό πλέον, αλλά αμοιβαιότητα, ισοτιμία στο εμπόριο, διότι οι δημόσιες προμήθειες δεν καλύπτονται τη συμφωνία GATT ή GATT. Οπότε, το άνοιγμα των αγορών για τις ευρωπαϊκές εταιρείες θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης και σε οικονομική ανάπτυξη. Ε, πιστεύω ότι η γνωμοδότηση αυτή αξίζει να υποστηριχθεί και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, και αυτές τις συζητήσεις με το Συμβούλιο. Είχα την ευκαιρία να τα συζητήσω σε διάφορες ε, ομάδες εργασίας της Επιτροπής μας με εκπροσώπους των κατώμελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας θα μπορούσε να μας ενημερώσει ε, για το ποιε χώρε εναντιώνονται στην πρόταση αυτή. Η δική μου χώρα, λόγου χάρη, νομίζω ότι είναι ενάντια. Αλλά ε, στο Συμβούλιο πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι κρίμα να μην ε, διαθετήσουμε αυτόν τον τομέα. Δεν θέλουμε να είμαστε προστατευτικοί. σα ίσα να έχουμε ισοτιμία στο εμπόριο με ισότιμη συμμετοχή εταιριών τρίτων χωρών στι δικέ μα δημόσιε προμήθειε και τούμπαλιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γκραπίνη. Και κυρία Μακλάκη, από του συντηρητικού μεταρρυθμιστέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή και μετά του συναδέλφου. Είχαμε πολύ επικοδομητική συνάντηση χθε. Στη συνάντησή μα καλωσορίζουμε τι τροπολογίε που έχουν υποβληθεί από τι υπόλοιπε ομάδε και ελπίζουμε να εργαστούμε σε ένα θετικό κλίμα όλοι μαζί για να βρούμε λύσει. Όπως καταστήσαμε σαφές, η δική μας ομάδα ε, συμμερίζεται το σκοπό και το στόχο να υπάρξει μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών και ε, αυτό για ευρωπαϊκές εταιρείες, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό είναι να απελευθερωθούν οι εμπορικές συμφωνίες και όχι με αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση αναγκαστικά. Ε, και δεν χρειάζεται να υπάρχει εργαλείο για το θέμα αυτό. Επίση, εκτιμούμε το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση έχει καταστήσει σαφέ ότι δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να κλείσει ε, τώρα η αγορά προμηθειών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Θα πρέπει να κοιτάξουμε μήπως εδώ με τα μέτρα αυτά δημιουργούνται περιπτώσεις αποκλειστικής αρμοδιότητας ε, και επηρεαστούν οι σχέσει μα με τρίτε χώρες. Εκεί μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει να άρει φραγμούς ε, συμμετοχή μα σε διάφορες δημοσίες προμήθειε. Αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο για μέτρα προστατευτισμού και περιορισμού των δυνατοτήτων μα. διότι πιστεύουμε ότι αυτό το είδου η πολιτική και αυτό το είδου το εργαλείο για το άνοιγμα των αγορών ε, μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίε αν εμεί άρουμε φραγμούς για άλλα κράτη στην δική μα αγορά. Θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο. Εάν υπάρχει εξαίρεση για τις μικρομεσαίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει το ίδιο να ισχύει και για δυνατότητα άλλων αγορών που μπορεί να ε, άρουν φραγμούς προστατευτισμού κατά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τη Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, φροντίσουμε να έχουν τη δυνατότητα οι μικρομεσαίε μα να έχουν πρόσβαση σε νέε αγορέ και αυτό το αντίστροφο. Θα πρέπει να φροντίσουμε, να διαχωρίσουμε τον προστατευτισμό από την προσπάθεια ανοίγματο και να φροντίσουμε να μην υπάρξει οπισθοχώρηση σε σχέση με την εμπορική απελευθέρωση που έχουμε πετύχει ω τώρα. Επίση, θα πρέπει να είμαστε εμεί παράδειγμα για του υπόλοιπου και να πω ότι διαφωνούμε ε, γιατί ε, σε σχέση με, το, με τη γνωμοδότηση που αποβάλλεται υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Εκεί συμφωνούμε λοιπόν με τον εισηγητή και μπορούμε να ε, παραμείνουμε στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, απο, Επιτροπής μας αποκλείοντας τροπολογίες που θα μπουν ε, και θα ε, παρέμβουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Αυτά πρέπει να τα δούμε από κοινού. Δεν θα στηρίζαμε καμία τροπολογία που θα ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει την επιβολή ε, περιορισμών στην αγορά δημοσίων προμηθειών. Δεν είναι εδώ το σημείο να γίνει αυτό και δεν θα συμφωνήσουμε με καμία τροπολογία που θέλουν ευρωπαϊκό νομοθέτημα για να, που μπορεί να υπονομεύει την αγορά των ε, προμηθειών και το οποιοδήποτε μέτρο προστατευτισμού. Αυτή είναι η άποψή μα ε, στου ιδρυτικού και μεταρρυθμιστέ. Θα συνεργαστούμε με τι άλλε ομάδε ε, για να το πετύχουμε, αλλά αυτό που θέλουμε ε, για να έχουν πρόσβαση μικρομεσαίε μα επιχειρήσει σε νέε αγορέ δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουμε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την Άλτε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του εξετάζοντας τις τροπολογίες για την Άλλοι για την ώρα δεν βρίσκω ε, πολύ κοινό έδαφος μεταξύ των σκιωδών. Μερικοί, ε, μερικές τροπολογίες δικαιολογούν ε, τον προστατευτισμό απέναντι στις τρίτες χώρες και η ομάδα μου δεν μπορεί να τις υποστηρίξει πρέπει να αγωνιστούμε κατά του προστατευτισμού και υπέρ του ελευθέρου εμπορίου, όπως είπε η Προεδρία η Εστονική. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε ε, τον προστατευτισμό όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίω. Κλείνοντας τις θύρες ε, θα οδηγηθούμε σε όλο και περισσότερες κλειστές θύρες και αυτό ε, θα βλάψει την ευρωπαϊκή οικονομία, της ευρωπαϊκής μικρομεσαίες επιχειρήσης. σχετικά βεβαίως, οι όροι οι κοινωνικοί δεν έχουν τίποτα να κάνουν με το στόχο του μέσου. Παρόλο που δεν ε, συμφωνούμε με το μέσο αυτό, η λογική του πρέπει να ε, γίνει σεβαστή. Ε, είχαμε την θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρώτη πρόταση. Θα θέλαμε ο εισηγητής να περιοριστεί στην αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής. Έχουμε επίσης τροπολογίες που προσπαθούν να ε, τροποποιήσουν ορισμούς που ήδη υπάρχουν ε, στην τομέα των δημοσίων συμβάσεων και δεν έχει κανένα νόημα να τροποποιούμε τον ορισμό αυτό για αυτό το μέσο. Η ομάδα μου θα υποστηρίξει ε, τις τροπολογίες του εισηγητή, αλλά δεν, δεν βλέπω που είναι οι συμβιβαστικές τροπολογίες αυτή. Νομίζω ότι ο εισηγητής θα πρέπει ε, να ψηφιστούν οι τροπολογίες μέσω των δυνατόν πιο ομαδικές ε, ψηφοφορίες. Ε, θα ψηφίσουμε για την απόρριψη της πρότασης που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει. Ελπίζω ότι ότι η Κομισιόν θα ασχοληθεί με την πρόταση. Η πρώτη εκδοχή δεν είναι αποδεκτή από το Συμβούλιο και από μένα. Δεν δεν βλέπω τις αλλαγές που απαιτούνται με την τροποποιημένη πρόταση. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο σκιώδη εισηγητή ή άλλο μέλος που να επιθυμεί να λάβει το λόγο. Θα επανέλθουμε λοιπόν στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Όχι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Η Επιτροπή επίσης θέλει να λάβει το λόγο. ο Ζων Ιβνόλερ από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε ε, την ε, ευκαιρία να αντιδράσω σύντομα, να απαντήσω κατά τη διάρκεια της ε, τελευταίας συνεδρίασης ΙΜΚΟ ε, μπόρεσα να αναφέρω την ανάγκη για ένα μέσο διεθνές για τις συμβάσεις δημοσίων αγορών για να ενισχύσουμε τις διεθνείς διαπραγματεύσεις ε, ξέρετε ότι είναι ανοιχτή αγορά δημοσίων συμβάσεων η ευρωπαϊκή, ενώ τα αγαθά μας και οι υπηρεσίες μας έχουν ε, εμπόδια σε τρίτες χώρες όπου υπάρχουν προτιμησιακά καθεστώτα, όπως η Κίνα, παρέντος χάρη. Και έχουμε και άλλους εμπορικούς εταίρους εκτός Ευρώπης. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στους εταίρους να επιφέρουν διακρίσεις ε, για τις ευρωπαϊκές αγορές, όταν οι δικές μας αγορές είναι ανοιχτέ στη διεθνή ανταγωνισμό. Ε, ε, χαιρετίζω την συζήτηση εδώ στην Επιτροπή και θα συζητήσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες που έχουν εκπονηθεί. Ε, θα χαιρετίζαμε κάθε επικοδομητική τροπολογία που θα διευκρίνιζε το πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής και την εφαρμογή του μέσου, ε, κυρίως για τις συμβάσεις παραχωρήσεως. Και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο ε, για τον κατάλογο των αρχών σχετικά με τις συμβάσεις αυτές, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι συνεκτικό με τον γενικό στόχο ε, της ενιαίας αγοράς. Υπάρχουν τροπολογίες που κατατέθηκαν ε, που σχετίζονται ε, με την θεμητό ανταγωνισμό. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι συμμεριζόμαστε την, την άποψη αυτή και αυτό λέχθηκε στην προηγούμενη οδηγία μας και πάλι εδώ είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για το σκοπό αυτό με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Θεωρούμε την πρόταση αυτή ως εξαιρετικά σημαντική και μας ενθαρρύνουν τα συμπερέσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που κάλεσε το Συμβούλιο και την Κομισιό να προωθήσει τη συζήτηση για το πώς να εξασφαλίσει αμοιβαιότητα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων για να υπάρξει και άλλη απόφαση στο Συμβούλιο σε συμφωνία με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο σε συζήτηση. Ε, θέλουμε να λάβουμε τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες και να συνεργαστούμε με τα μέλη του Κοινοβουλίου για να βελτιώσουμε το κείμενο της πρότασης της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στεφανέκο, εισήγητης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι η ιστορία του θέματος είναι ενδιαφέρουσα, το ιστόλο ιστορικό και υπάρχουν διάφορες θέσεις από διάφορες ομάδες. Θα προσπαθήσω να βρω μερικά συμβιβασμούς και κοινό έδαφος και χαίρομαι που περίπου όλοι ενδιαφέρονται για μια κοινή θέση. Θα προσπαθώ όσο το δυνατόν καλύτερα να επιτύχω συμβιβαστικές λύσεις ούτως ώστε να προχωρήσουμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και καλή τύχη. Ε, στις 25 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην ΙΜΚΟ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο χρόνο για την επόμενη συζήτηση που είναι σημαντική συζήτηση επίκαιρη που θα έχουμε τώρα τα προϊόντα οικοδομών, τον κανονισμό και την ασφάλεια, την πυρασφάλεια. Και η ε, Κάτριν Στίλερ είναι η συγγήτρια και όλοι ξέρουμε γιατί το θέμα αυτό ενέχει τόσο μεγάλη σημασία λόγω ε, της ε, πυρκαγιάς στο Γκράνφελ Τάουερ και αυτή η ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποβλέπει την ε, συζήτηση σχετικά με τον κανονισμό για τα οικοδομικά υλικά, ναι. ε, την ενδεχόμενη αναθεώρηση ε, του κανονισμού και το πώς σχετίζεται με την πυρασφάλεια. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα μπορούσε να περιλάβει βεβαίως ε, μια ε, παρουσίαση πρωτοβουλειών που έχουν αναλυφθεί σχετικά με το θέμα αυτό. Άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που έβαλε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, το που είναι σημαντικό για μας τους νομοθέτες να έχουμε αυτές τις συζητήσεις για επίκαιρα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες. Γι' αυτό χαίρομαι που σου δίνω το λόγο. Κύριε Στάιλερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που υποστηρίζετε αυτή την πρωτοβουλία σήμερα. Όλοι με φρίκη και τρόμο είδαμε τι συνέβη στο Λονδίνο και ανέκυψαν πολλά ερωτηματικά ως προς την πύρα, ασφάλεια των οικοδομικών υλικών και ποιος έχει την ευθύνη. Εμείς έχουμε ευθύνη για τον κανονισμό που διέπει τα προϊόντα τα οικοδομικά υλικά και καλό είναι να το σκεφτούμε, να προβληματιστούμε και να δούμε τι δράσεις μπορούμε να αναλάβουμε. Για να είμαστε σαφείς, εδώ δεν πρόκειται για απαιτήσει για τα οικοδομικά υλικά, αλλά για εναρμόνιση των κανόνων και πώς ε, θα έχουμε το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CE, και τι εγγυάται αυτό τα ενεργειακά, τα περιβαλλοντικά τα ορίζουν τα κράτη-μέλη ως πρότυπα. Γι' αυτό έχει κάποια περιπλοκότητα το θέμα. Υπάρχουν ε, διάφορα ζητήματα που ανέκυψαν, όχι μόνο για την αναθεώρηση του ίδιου του κανονισμού, αλλά γίνονται και συζητήσεις ε, για τις προσώψεις των κτηρίων. Ε, ξέρουμε σε σχέση με την ε, πυρκαγιά στον ε, πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου. Ξέρω ότι παρευρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μας ενημερώσει για τα θέματα αυτά. Αλλά τι γίνεται με τις προσώψεις, τις επικαλύψεις, τα κτίρια. Και είναι ενδιαφέρον να ακούει κανείς ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν σαφείς κανόνες για το πώς χρησιμοποιούνται πια υλικά, ενώ σε άλλες χώρες όχι. Αυτό εναπόκειται στην κάθε χώρα, δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, το ξέρω. Αλλά αυτά τα θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν και να τα κοιτάξουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια γενικότερα ζητήματα πύρα ασφάλειας. Δεν είχαμε στρατηγική από το 1986. Οπότε ε, νομίζω ότι χωράει κάποια δράση εδώ. Και πάλι αυτό έχει να κάνει ε, γενικότερα, όχι με το συγκεκριμένο κανονισμό για τα οικοδομικά υλικά. Ε, πώς θα ε, καθορίσουμε μια στρατηγική. Το άλλο που έχει να κάνει με τον κανονισμό όμως για τα οικοδομικά υλικά είναι η τοξικότητα. Είναι ποσοτικό το ζήτημα, η λύση δεν είναι εύκολη. Υπάρχει διεθνές πρότυπο για την τοξικότητα. Δοκιμάζονται αυτά τα πράγματα, ελέγχονται, εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είναι τα ερωτήματα και πολλά. Τι θα κάνουμε τον κανονισμό για τα οικοδομικά υλικά, τι γίνεται με την τοξικότητα, μπορούμε να έχουμε καλύτερους κανόνες σχετικά, τι γίνεται για την τρέχουσα ε, μεταρρύθμιση των υλικών που χρησιμοποιούνται στις προσώψεις και γενικότερα πώς αντιμετωπίζουμε την πυρασφάλεια. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία γιατί έχουμε από τη μια τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και πρέπει να δούμε πού μπορούμε να μοιραστούμε τις καλές και τις βέλτιστες πρακτικές για να έχουμε προστιθέμενη αξία αλλά και να διδασκόμαστε ένα από τον άλλον. Όλα αυτά λοιπόν μα οδήγησαν στο να γράψουμε το σημείο αυτό στη μέση διάταξη. Ξέρουμε ότι στις 13 Σεπτεμβρίου θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια. Παρακαλώ σημειώστε το, τρει ώρα το μεσημέρι προβλέπετε για το Στρασβούργο. Παρακαλώ ελάτε και, ελπίζω, και χαίρομαι που έχουμε εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ξέρω, είναι και θέμα των κρατών μελών. Το συζητήσαμε και με την Εστονική Προεδρία το πρωί. Και το είπαμε στις υπουργού ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει και τα κράτη-μέλη να προβληματιστούν και να κάνουν προτάσεις για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ελπίζω, Πρόεδρε, να βοηθήσει αυτό ως εισαγωγή θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί τώρα ενδιαφέρει τους πολίτες και έχουμε και κάποια ευθύνη λόγω του κανονισμού για τα οικοδομικά υλικά. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα. Χαίρομαι που βλέπω παρόντες τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται και θέλω να παρακαλέσω και το ε, Κομισιόν και την Εστονική Προεδρία ενδεχομένω να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Κάθριν. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσω το λόγο στην κυρία Φούλβια Ραφαέλη ε, από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστώ κυρία Στήλερ για την εισαγωγή και για το ότι βάλατε το θέμα στην ημερήσια διάταξη μετά την πυρκαγιά στο Grenfell ε, Tower το θέμα αυτό έχει τεθεί, είναι επίκαιρο θέμα, συζητείτε πολύ και είμαι εδώ για να σας ε, πω ποια είναι η προσέγγιση μας σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο επίπεδο των κρατών μελών και ποια είναι τα μέτρα που η Κομισιόν έχει ήδη λάβει και ε, προτίθεται να λάβει για αυτά τα θέματα ασφαλείας με τις διατάξεις της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την ασφάλεια των κτηρίων για τους πολίτες. Είναι αδιάψευστο γεγονός ότι οι διαφορές, οι κλιματικές, οι γεωγραφικές υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών ε, σχετικά με την σεισμικότητα, με την χρήση διαφόρων υλικών ε, οικοδομικών. Ε, ίσως σε επίπεδο κρατών μελών η ασφάλεια εξασφαλίζεται καλύτερο και μέχρι τώρα η Κομισιόν δεν ε, διαθέτει ε, την γνώση ότι οι διατάξεις εθνικές δεν είναι επαρκής. Χρειαζόμαστε καλύτερα ενεργειακά κτίρια σε σχέση με το, τα κτίρια που υπάρχουν και, και έχουμε μεγάλη επιλογή προϊόντων που προσφέρονται στην αγορά δύο πράξεις είναι αποφασιστικές σχετικές με τις ανάγκες μετά την καταστροφή αυτή. Πρώτα έχουμε τον κανονισμό για τα οικοδομικά ε, υλικά και την οδηγία για την ενέργεια. Θα μιλήσω για τον κανονισμό σχετικά, το CPR, τον κανονισμό για τα οικοδομικά προϊόντα. Ο κανονισμός αυτός το 2011 όπως είναι σήμερα η νομική βάση 114 της συνθήκης και ο στόχος του κανονισμού είναι να ενοποιήσει την αγορά για τα οικοδομικά υλικά με κοινού κανόνες σχετικά με τα πώς θα αξιολογούνται οι αποδόσεις ε, από τους κατασκευαστές των προϊόντων. Τα κράτη-μέλη έχουν λοιπόν την αρμοδιότητα να ρυθμίζουν την ασφάλεια με απαιτήσει σχετικά με την απόδοση των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στα κτίρια όταν θεωρούν ότι αυτό είναι κατάλληλο χάρη, τα, οι αρχές των κρατών μελών μπορούν να αποφασίσουν ε, αν τα προϊόντα τα τα που δεν καίγονται είναι κατάλληλα ή όχι. Η, το πρότυπο του, του κανονισμού CPR ε, λέει απλώς πώς να αξιολογεί κανείς ικανοποιητικά τις αποδόσεις και πώς να τις κοινοποιεί. Θα ήθελα τώρα να εξηγήσω και να διευκρινίσω ε, κάτι το οποίο έχει σχέση με τα οικοδομικά προϊόντα. Τα οικοδομικά προϊόντα έχουν ένα σήμα. Αλλά το σήμα αυτό δεν δείχνει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις οικοδομικές εργασίες. Αυτό το σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι ο κατασκευαστής του προϊόντος έχει δηλώσει ε, την απόδοσή του σε σχέση με βάση τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά τα αντίστοιχα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κτίριο που χρησιμοποιείται το προϊόν είναι ασφαλές. Αυτό καθορίζεται από κανονισμό εθνικό του κάθε κράτους μέλους. Από όλα τα προϊόντα με σήμα, μόνον αυτά που έχουν την απόδοση που απαιτείται από τον ε, κανονισμό ε, ε, κατασκευής, οικοδόμησης και κτηρίου. Αυτή είναι σημαντική διαφορά ανάμεσα στον κανονισμό CPR και άλλες νέες νομοθεσίες πλαισίου όπως την οδηγία περί μηχανημάτων. Βάσει του CPR τα καλύπτεται το ότι ασφάλεια υπηρασφάλεια είναι η αντίδραση στην πυρκαγιά των προϊόντων, η αντίσταση, η ανθεκτικότητα των προϊόντων και η, πόσο στεγανά είναι στην πυρκαγιά. Αυτά έχουμε κατηγορίες επιδόσεων και μέθοδους ελέγχου για τα προϊόντα τα οικοδομικά. Ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από την νομοθεσία είναι αυτά που δεν αντέχουν στην πυρκαγιά και αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υπηρεσίες έχει ε, δώσει εντολή για δύο μελέτες ε, για αυτές τις απόψεις. Η πρώτη μελέτη σχετικά με την τοξικότητα του καπνού για να ελέγχεται η τοξικότητα από, που προέρχεται από το προϊόντα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μέχρι τώρα η Κομισιόν δεν διαθέτει αποδείξεις ότι τα κράτη-μέλη έχουν ρυθμίσεις για το θέμα αυτό. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ελλείψεις των ρυθμιστικών ε, προσεγγίσεων της τοξικότητας ε, του καπνού σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων αν ε, συγκριθούν με προληπτικά μέτρα όπως συναγερμό, πυρκαγιάς κλπ. Αυτό υποστηρίζεται από διαπιστώσεις ότι ίσως ε, η πυρκαγιά διαδίδεται από το περιεχόμενο του κτηρίου και όχι από τον ε, καπνό, η τοξικότητα που προέρχεται από τη φωτιά έχουμε την παρακολούθηση μετά την μελέτη και θα δούμε τι συνέχεια θα δοθεί στην μελέτη αυτή. Η δεύτερη μελέτη που, ε, που το 2016 ζητήθηκε από την Κομισιόν η Ευρωπαϊκή ε, Προσέγγιση για την αξιολόγηση της πυρκαγιάς. Το σημείο εκκίνησης της μελέτης είναι μια προσέγγιση που περιλαμβάνει ελέγχους ε, όχι μόνο σε μεγάλο βαθμό αλλά και σε μικρή κλίμακα διότι μερικά κράτη-μέλη παρουσιάζουν ε, ότι, ότι χρησιμοποιούν μέτρα και οι αρχές δεν θέλουν να εγκαταλείψουν αυτήν την προσέγγιση. Η ασφάλεια δεν, ε, ε, δεν εξαρτάται μόνο από την πρόσωψη και ακόμα και αν υπάρχουν έλεγχοι μεγάλης κλίμακος μπορεί να υπάρξει τέτοιος κίνδυνος. Στον φθινόπερο θα ξανασυζητήσει η Κομισιό με όλα τα κράτη-μέλη την ανάγκη να διατηρηθούν ε, σε αυτήν την προσέγγιση αξιολόγησης ε, μικρής κλίμακας έλεγχη και οι ρυθμιστές ε, είναι έτοιμοι να δεχθούν ίσως μόνο τα μεγάλης κλίμακος. Η μελέτη για την τοξικότητα καπνού θα δώσει για τα, όχι μόνο για την Κομισιό αλλά και για τα κράτη-μέλη στοιχεία ούτω ώστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Το δεύτερη νομοθετική πράξη που συζητείται πολύ μετά το Grenfell, PB, που απαιτεί τα κράτη-μέλη ε, στις κώδικες ε, τους εθνικούς να έχουν ελάχιστες απαιτήσεις στο Διεθνές Κώδικα Κτηρίων ε, για την ε, θερμική απόδοση σχετική, ε, σχετική με τους τείχους, με τις ορεφείς, για τα συστήματα ψήξης και έχουμε τις διεθνείς κανόνες. Η PBD δεν έχει απαιτήσει σχετικά με την απόδοση των οικοδομικών υλικών. Δεν έχει λοιπόν επίδραση στην στην απόδοση των προσώψεων. Σχετικά με τα οικοδομικά υλικά ε, έχουμε, είναι θέμα επικουρικότητας. Σχετικά με τις απαιτήσει εθνικές, το EPB δεν ασχολείται με ε, τα με τις χαρακτηριστικά των υλικών και το ε, γενικό πλαίσιο για την ενεργειακή αποδοτικότητα δεν λαμβάνει υπόψη τις εθνικές απαιτήσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα μέτρα που απαιτούνται για ε, τα οικοδομικά υλικά για να υπάρξει μεγαλύτερη πυρασφάλεια που να οφείλεται στα υλικά, όπως ξέρετε, οι ε, κανονισμοί σήμερα ε, είναι θέμα εφαρμογής από τις αρχές των κρατών μελών και για την ώρα δεν έχουμε καμιά απόδειξη ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι έλεγχοι σε εθνικό επίπεδο. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες ε, σχετικά ε, για το, με το θέμα του Grenfell Tower. Σε αυτή τη στιγμή ε, η πυρκαγιά αυτή οδηγεί σε διάφορα ερωτηματικά σχετικά με την εξωτερική θερμική μόνωση του κτηρίου και με εσωτερικά θέματα και θα πρέπει να ε, έχουμε διάφορες γνώσεις συμπληρωματικές για την πυρασφάλεια. Τα κράτη-μέλη έχουν δύσκολη πρόκληση σχετικά με το θέμα. Τα, τα κτίρια ε, και η ασφάλειά τους δεν οφείλεται μόνο ε, στα υλικά, οφείλονται και στο σχεδιασμό, σχεδιασμός, η συντήρηση των συστημάτων συνεργερμού, πυρασφάλειας και εξαρτώνται ε, η ασφάλεια του κτηρίου εξαρτάται από πάρα πολλά στοιχεία. Τα θύματα τα 30 τελευταία χρόνια είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και ε, και οφείλεται ο θάνατός τους σε απορρόφηση διαφόρων αερίων, σε εισπνοή διαφόρων αερίων στην αρχική φάση της πυρκαγιάς όταν οι άνθρωποι θα μπορούσαν να επιζήσουν πάρα πολλά κράτη-μέλη ζητούν την κατάλληλη εφαρμογή τέτοιων διατάξεων, αλλά αυτές οι διατάξεις εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη. Η Κομισιό είναι έτοιμη να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στις αναλύσεις τους και έτοιμη να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ε, των αντιστοίχων ε, εθνικών αρχών και των ενδιαφερομένων ούτω ώστε να μάθουν ποιες είναι οι βαλτίστες πρακτικές όσον αφορά την ε, οικοδημικά υλικά και την ε, κατασκευή. Νομίζω ότι αυτό θα ενισχύσει την ικανότητα των κρατών μελών και των ρυθμιστικών αρχών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους γνωρίζοντας καλά τις ε, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επιλογών τους. Ευχαριστώ για την προσοχή. Thank you very much for this... Σας ευχαριστούμε για αυτή την εμπεριστατωμένη ενημέρωση. Θα ζητήσω τώρα από του υπόλοιπου συναντέλφου που θέλουν το λόγο ή να θέσουν ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνουν. Ο κύριο Φαμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Κάθριν Στάιλερ που ως προεδρή συγγήτρια για τον κανονισμό για τα οικοδομικά υλικά μας έθεσε υπόψη αυτό το θέμα. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ισόρροπη πραγματικά παρουσίαση. Δύο σημαντικά θέματα έχω να αναφέρω. Πρώτον, βεβαίως είναι σημαντικό μετά από αυτό το φρικτό δυστύχημα στο Λονδίνο να δούμε κατά πόσο οι προδιαγραφές έφτεγαν ή η πλημελής ανάθεση ή πλημελής εκτέλεση ε, κάποιων διατάξεων ευθύνονται για αυτό το φρικτό ε, δυστύχημα. Πρέπει όμως αυτό να εξεταστεί σε βάθος. Και έτσι κατάλαβα εγώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση και δεν πρόκειται να εξυπηρετήσουμε κανένα όταν κάνουμε χάρη σε κανέναν ε, εάν τώρα σπεύσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Θα πρέπει σε βάθος να μελετηθεί και να ελεγχθεί. Βεβαίως και είμαι υπέρ αυτού και ευχαριστώ για τις ε, προτάσεις. Θα δούμε τα συμπεράσματα αργότερα. Έμαθα ε, πώς χτίζονται κανονικά ε, και πώς εξοπλίζονται τέτοια κτίρια. Στη Γερμανία από 22 μέτρα και πάνω πολυκατοικίες έχουν ειδικέ διατάξεις, εξωτερική τύχη και η επένδυσή τους πρέπει να είναι αποκλειστικά από πυρήμαχα υλικά. Αυτά είναι μεν εθνικές ρυθμίσεις, αλλά και άλλα κράτη-μέλη μπορούν να τα υιοθετήσουν. Και υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις που δεν θέλω να τις διαβάσω όχι και διατάξεις, αλλά και μόνο από μια επισκόπηση που έχω κάνει δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση ότι αυτό έχει να κάνει με τη σύνθεση ε, της μόνωσης της πρόσωψης, αλλά κυρίως με το πώς έχει ε, χτιστεί και εξοπλιστεί το κτίριο. Λοιπόν, θα ήθελα να προσθέσω ένα δεύτερο σημείο. Ακόμα και αν είχαμε αυτό το φρικτό δυστύχημα στο Λονδίνο, στον ε, πύργο Γκρέμφελ και ε, την ευθύνη που έχουμε να το ξεκαθαρίσουμε για τα θύματα, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει σφοδρός ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων κατασκευαστών μονοτικών υλικών στην Ευρώπη και δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει ε, στο να ε, αποκομίσει ένα πλεονέκτημα η μία πλευρά λόγω της πυρκαγιάς του Λονδίνου, πόσο μάλλον όταν δεν έχει διαλευκανθεί ακόμα τι συνέβη. Παρακαλώ να κοιτάξουμε τα γεγονότα, τα πραγματικά στοιχεία και από εκεί και πέρα βγάλουμε συμπεράσματα και όχι αντίστροφα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι συμφωνούμε σε αυτό, οπότε προσβλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον στη συνέχεια αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Thank you very much. And then, uh, please. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σάλτεμόζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Στάιλερ που ε, οργάνωσε αυτή τη συζήτηση. Είναι σημαντικό να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αντιλήσουμε διδάγματα από αυτή την τραγική ε, υπόθεση στο Λονδίνο. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διεξοδικά μας παρουσίασε τους κανόνες ή την έλλειψη κανόνων ε, που αφορούν την ανάληψη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί τελικά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Έχω δύο σχόλια ουσιαστικά. Είμαι ευρωβουλευτής εδώ και 10 χρόνια. Θα πω ότι έχω μιλήσει επανειλημμένως με πυροσβέστες από όλη την Ευρώπη που θα ήθελαν να κάνουμε περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να προστατεύσουμε τις εργασιακές του συνθήκες και το δικό τους εργασιακό περιβάλλον. Νομίζω ότι και αυτό καλό θα ήταν να το έχουμε υπόψη, διότι η τοξικότητα των ε, αερίων είναι αυτό που ανησυχεί τους πυροσβέστες. Ε, να ακούσουμε εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν για τα τεστ τοξικότητας του υλικού που χρησιμοποιείται για πυρόσβεση οι πυροσβέστε λένε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να προστατεύονται και εκείνοι και πρέπει να τους ακούσουμε. Και το άλλο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι η ασφάλεια από τις πυρκαγιές, η προστασία από τις πυρκαγιές είναι θέμα και εθνική αρμοδιότητα, είναι θέμα των κρατομελών και εθνική αρμοδιότητα. Όμως πρέπει να βεβαιωθούμε για την προστασία των πολιτών με καλύτερη ίσως δειγματοληψία, συγκριτική αξιολόγηση με καλύτερο σύστημα καταγραφή των αναγκών του. Εάν κανεί ζει σε έναν ουρανοξύστη ε, σε μια οποιαδήποτε χώρα τη Ευρώπη, δεν πρέπει να γνωρίζει ποιε είναι οι προδιαγραφέ για την προστασία από πυρκαγιέ ε, στη χώρα του. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες, ενημέρωση για τους πολίτες, για την προστασία από πυρκαγιές σε αυτό το τομέα. Ξέρω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, καλά κάνετε, αλλά κάντε περισσότερα κατά περισσότερο ό,τι αφορά την ε, προσφορά δυνατοτήτων στα κατεμέλια για να ανταλλάξουν εμπειρίε. Πιστεύω πάντω. Ε, πιστεύω ότι οι πολίτες ε, μπορούν να μάθουν από την ανταλλαγή καλών εμπειριών μεταξύ τους δεν είναι ακόμα ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αλλά εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να, μπορεί να μας βοηθήσει τουλάχιστον να μοιραστούμε σωστά τις γνώσεις για να γνωρίζουμε τι είναι επιτυχημένο και τι όχι. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την πρόληψη των ε, τεράστιων καταστροφών όπως αυτή που είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες στο Λονδίνο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Κάθριν που έγραψε το θέμα αυτό στη Μέση Διάταξη. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να το συζητούμε. Κοιτάξτε, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να αποφανθεί η έρευνα τι συνέβη, το πώς και το γιατί. Συνέβη και ήταν τόσο ολέθριο αυτό το δυστύχημα στο Βεγκρέμφελ. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι το 60% της μείωσης από πυρκαγιές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι καλό, αλλά όταν βλέπεις μια τέτοια τραγωδία ο, ο κόσμος έχει δίκιο που μας λέει ότι δεν αρκούν όλα αυτά και φυσικά δεν αρκούν. Ξέρω ότι έχουμε περιορισμένο ρόλο εδώ όλοι μας, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τα κράτη-μέλη και ερωτηματικά. Ε, εξ όσων γνωρίζω, ε, αυτή η μόνωση που έχει μπει στην πρόσωψη ε, απαγορεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία και αλλού και μπορεί να είναι απαγορευμένη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, δεν το ξέρουμε ακόμα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγα μπορεί να κάνει, περιορισμένα πράγματα. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε κατά τη γνώμη μου. Και υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Εδώ εστιάζουμε λίγο στην τοξικότητα, που και αυτό είναι πολύ σημαντική. Αλλά συγκεκριμένη περίπτωση γνωρίζουμε ότι η ίδια η μόνωση, το υλικό οδήγησε στο να επεκταθεί η πυρκαγιά και να είναι η φωτιά πολύ χειρότερη από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Μην κοιτάμε μόνο την τοξικότητα των αερίων ε, της καύσης, που αυτό φυσικά είναι το πιο επικίνδυνο, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η ταχύτητα διάδοση φωτιάς λόγω του υλικού. Έχω λοιπόν ερωτήσεις γενικότερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασμό κτηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε υψηλά πρότυπα παντού γιατί ε, αυτό έχει να κάνει και με το σχεδιασμό του κτηρίου, όχι μόνο του συγκεκριμένου. Πολλά είναι τα κτίρια ανά την Ευρώπη που έχουν αμφισβητούμενη σχεδίαση ω προς την ασφάλειά τους. Και μετά κάποιες από τις βελτιώσεις που μα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πόσο χρόνο νομίζετε θα χρειαστεί για να υλοποιηθούν, όπω μέθοδοι δοκιμών και ο έλεγχος τη ασφάλειας, ως προς την τοξικότητα των υλικών γιατί έχουμε κάνει πολλή δουλειά σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ και πάλι Κάθριν που ανακοίνησε σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος. Υπάρχει άλλος βουλευτής που να θέλει να μιλήσει, που να είναι παρόν. Όλα αυτά που ήθελα να πω εγώ υπόθηκαν, με καλύψατε. Ευχαριστώ την Κάθριν που ζήτησε να εγγραφεί το θέμα στην ημερησία διάταξη. Την ε, ευχαριστώ και προηγουμένως για να μας απαντήσει παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Συμφωνώ απολύτως ότι ακόμα και ένας νεκρός από πυρκαγιά είναι υπερβολικός αριθμός θυμάτων αλίμονο. Δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα. Δεν πρόκειται για ζωές. Συμφωνούμε ότι πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές στα κράτη-μέλη και όντως αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να δημιουργήσει αυτή την πλατφόρμα. Θα πρέπει να το συζητήσουμε και με το Συμβούλιο και με την Προεδρία, διότι πραγματικά αυτό είναι θέμα των κρατών μελών. Δεν χωράει καμία αμφιβολία θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε και να βελτιώσουμε τα πράγματα γιατί ε, υπάρχει προστιθέμενη αξία. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις έγιναν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενημέρωση για τέτοια έγγραφα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να το διερευνήσουμε ε, βάσει των ε, βελτίστων πρακτικών δεν ξέρω, χρειάζονται έγγραφα κοινή αναφορά, κοινών προδιαγραφών, ένα κοινό σύστημα αναφορά. Θα το μελετήσουμε, γιατί όχι. Σε ό,τι αφορά τι μελέτε, ιδιαίτερα τη μία ε, μελέτη για την τοξικότητα των ε, καπνών, των αερίων, τον φθινόπωρο θα ε, ολοκληρωθεί η μελέτη και θα δούμε τι δράσεις μπορούμε να αναλάβουμε βάσει της μελέτης αυτής. Και πάλι θα δούμε αν χρειάζεται ένα πρότυπο για να ε, γίνονται οι δοκιμές και οι έλεγχοι τοξικότητας του καπνού από την καύση των οικοδομικών υλικών. Υπάρχει ο κανονισμός για τα οικοδομικά προϊόντα. Δεν είπα ότι αναθεωρείται αυτός ο κανονισμός αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό έχει ξεκινήσει πολύ πριν το δυστύχημα και δεν έχει άμεση σχέση με ζητήματα πυρασφάλειας. Τώρα θα ε, προκηρύξουμε μια μελέτη για τη ε, μελέτη του αντικτύπου ακριβώ και του κινδύνου. Αν χρειάζεται αναθεώρηση και ο κανονισμός αυτός. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κάθριν, δεν ξέρω αν θέλεις να έχεις το τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Νομίζω το ζήτημα που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι που το κοιτάζουμε τώρα. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κατομελών στις ε, δοκιμές και τα τεστ, μικρότερα, μεγαλύτερα. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Και το είπε και ο Άντριου. Η... Οι προσώψεις και η μόνοσή τους είναι ένα θέμα. Το είπε και ο Ανδρέας για το ε, τι ε, επίπεδου είναι τα πρότυπα. Επίσης, οι δοκιμές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανταλλαγή των πρακτικών, με την ανταλλαγή των δεδομένων είναι πολύ σημαντική για να ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε. Επίσης, το να κατανοούμε τους κανόνες για την προστασία από τις πρικαγιές στα διάφορα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό. Σε πολλά κράτη-μέλη, όταν ξεκινά μια πυρκαγιά, δίνονται τόσα λεπτά, δύο ας πούμε, για την ε, ειδοποίηση που ε, χρειάζεται. Σε κάποια άλλα κράτη προβλέπεται ένα δεκάλεπτο. Ε, αυτό έχει να κάνει με το τι υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των κτηρίων και είναι σημαντικό να κατανοούμε τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και πώς αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά, τις φωτιές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μπορεί να τα συγκεντρώνει σε μια πλατφόρμα, αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει να το φοδοτούν αυτή την πλατφόρμα. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην όλη προσπάθεια ε, υπεύθυνα. Το είπε και η κυρία Σάλτε για την τοξικότητα και κυρίως το τι συμβαίνει με τους ε, πυροσβέστες μας στα διάφορα κράτη-μέλη. Όταν υπάρχει μια φωτιά από ένα λατωματικό ψυγείο και δεν αντιμετωπίζεται Και επειδή έζησα την ιστορία αυτή με τους πυροσβέστες που το αντιμετώπισαν και μας είπαν πόσο γρήγορα απλώθηκε η φωτιά. Πρέπει να στηρίξουμε τους πυροσβέστες και να βεβαιωθούμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το θέμα εδώ είναι ότι είναι πολλοί οι πυροσβέστες προς την υγεία τους και το τι εμπειρίες έχουν ζήσει είναι κάτι που να το σκεφτούμε. Διότι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για την τοξικότητα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα κτίρια και όλα αυτά τα ζητήματα, Εάν μπορούμε να το σκεφτούμε και έχουμε κάποια ευθύνη ε, ή τέλο πάντων κάποια αρμοδιότητα για τα πρότυπα, να το κάνουμε και επίση, η γενικότερη στρατηγική μα για την προστασία από τι πυρκαγιέ. Εντάξει, για τα κτίρια και την ασφάλειά του είναι ένα θέμα που το εξετάζουμε τώρα, αλλά για μια ενιαία στρατηγική για τις πυρκαγιέ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολύ καιρό δεν έχουμε κάνει τίποτα. Από το 86 νομίζω ήταν η τελευταία πρωτοβουλία. Είναι λοιπόν κάτι που θα μπορούσαμε συνολικά να το σκεφτούμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι η πλατφόρμα είναι μια πολύ καλή αρχή και θα πρέπει να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι προσπαθίε τη. Αλλά θα πρέπει να ζητήσουμε και από τα κάτι μέλη να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι διαρκώ βλέπουμε ε, ότι αυτά τα πράγματα ε, είναι πολύ καλά γνωστά στα διάφορα ξεχωριστά, αλλά θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να τα σκεντρώσουμε και να τα μοιράζονται. Ευχαριστώ πολύ, Κάθριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Μπορούμε να πούμε ότι καλά κάναμε και γράψαμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και ήδη έχουμε και αποτέλεσμα να πρώτα αυτή την πλατφόρμα που προτείνουμε και να το διαδώσουμε και στα κράτη-μέλη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθατε. Άρα εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίαση της Επιτροπής μας για σήμερα. Η επόμενη συνεδρίαση θα είναι αύριο στις 9.30 για τις ψηφοφορίες και μετά θα πάμε διακοπές. Σας ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς. Οι διερμηνείς ευχαριστούν την Πρόεδρο και τη Γραμματεία για την προετοιμασία της σημερινής συνεδρίασης συντονιστές στη συνέχεια σε ένα τέταρτο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας.